στους συνεργάτες μας και την Ίγκε και τον Αλεσάνδρο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσά κύριε Δανέλη και επομένως τώρα θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Έκθεση Λουί Μισελ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό ε, για θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Παρακαλώ με την ησυχία σας. Κύριε Ντεκεζέρ, γρήγορα να προλάβετε να ψηφίσετε. Άψογα, πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Μισελ. Ψηφίζουμε τώρα την ε, έκθεση Μορέιδα Δυνατάσεως της Χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγκεκριμένα. Ε, η δεύτερη έκθεση Μορέιρα διονομαστικής κλίσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Υπερψηφίζεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια ε, κύριε Μορέιρα. Τρίτη έκθεση Μορέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εδώ έχουμε πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια για μια τρίτη φορά, κυρία Μορέιρα. Ε, σύσταση Σίμψον, διανατάσεως της χειρός, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια, κύριε Σίμψον. Επίσης, ε, έκθεση Σίμψον, μνημόνια συνεργασίας, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία για μία ακόμα φορά συγχαρητήρια. Τώρα, ε, δεν υπάρχουν τροπολογίες όσον αφορά τη, τα μέλη των επιτροπών. Ε, συμφωνούν όλοι. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Έκθεση Florence. Πρώτο μπλοκ, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. <clears throat> Πέρας. Εγκρίνεται. Γίνεται δεκτή λοιπόν η τροποποιημένη θέση του Συμβουλίου. Συγχαρητήρια κύριε Φλόρενς. Έκθεση Κρίστα Κλάς. Έχουμε δύο ομάδες τροπολογιών. Διονομαστικής κλήσεως η πρώτη ομάδα άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Γίνεται δεκτή λοιπόν η τροποποιημένη θέση του Συμβουλίου. Συγχαρητήρια κυρία Κλάς. Έκθεση Μποβέ. Παράγραφος 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε η επαλήθευση ή άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίσαμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος για τις ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Μα Μα είναι μετά αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή Ακούστε με λίγο. Ψηφίζουμε την παράγραφο 26 σε δύο τμήματα. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 31. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές Ε, παρακαλώ να επαληθεύσουμε. 42, παράγραφος 42, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 11, υπέρ. Να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. F λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Μποβέ ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Παρακαλώ. Ναι, μετά την έγκριση του κειμένου πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι έγινε μια συλλογική εργασία από όλη την Επιτροπή Γεωργίας και χάρη ακριβώ αυτή τη συλλογική εργασία μπορέσαμε να ασκήσουμε πιο έντονη πίεση στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ούτε ώστε επιτέλους στην Ευρώπη οι καλλιεργητές να λαμβάνονται υπόψη ε, όσον αφορά το κόστος και τα έσοδά τους. Και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με επέτρεψαν να εκπονήσω αυτή την έκθεση και συγκεκριμένα τον κύριο Λόρεντσεν. Ευχαριστώ κύριε Μποβέ. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Γιατί δεν θα προλάβουμε τροπολογία ένα. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Διανομαστικής κλήσεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6, διονομαστική ως άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία 4. Με τον ίδιο τρόπο άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Κοινή πρόταση ψηφίσματος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια. Έκθεση Πατριτσέλο. Παρακαλώ. Θέλει κάποιος να μιλήσει. Όχι. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Θα ήθελα να πω ότι ως προς το ψήφισμα αυτό για την ανισορροπία στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων, καλώ τους συναδέλφους από την Επιτροπή Άγκρη στο μέλλον να συνεργάζονται καλύτερα με εμάς τους υπόλοιπους, με τα μέλη της Επιτροπής δηλαδή για την εσωτερική αγορά και τον καταναλωτή, γιατί οι ίδιες ανησυχίες μας αποσχολούν. Επιθυμούμε εμείς να συγκεντρώσουμε τη δυνάμεις μας μαζί με εσά, να μην δουλεύετε γραφειοκρατικά, να έχουμε ένα πιο αξιόπιστα αξιόπιστο μήνυμα προς τον έξω κόσμο, κάτι το οποίο θα αυξήσει την αξιοπιστία μας γενικότερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη συνεργασία. Ναι, ε, φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι από την ε, Επιτροπή Γεωργίας θέλουν την συνεργασία με τις άλλες επιτροπές, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Προ, ε, λοιπόν, έκθεση Πατριτσέλο υπέρ, κατά, της πρότασης ψηφίσματος. Αποχές εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Πατριτσέλο. Έκθεση Καρόνα. Έκθεση Σαλβατόρε Καρόνα. Αποφυγή πατάλης τροφίμων. Παράγραφος 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 28. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Καρόνα. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη. Επεξηγήσεις ψήφου λοιπόν επί των ε, συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άννα.